θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στο χθεσινό εσεμινάριο. Και όσους συμμετέσχουν και όσους είχαν την καλοσύνη να εισηγηθούν των τεσσάρων θεμάτων και να βγάλουν και τα συμπεράσματα. Θα επανέλθουμε, θα κάνουμε δηλαδή την briefing και μαζί θα δούμε τις κύριες γραμμές που πρέπει να εμβαθύνουμε για να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική η δουλειά μας. Τώρα δεχτείτε παρακαλώ μια τροποποιησούλα της ημερήσιας διάταξης και στις ψηφοφορίες να ψηφίσουμε πρώτα την έκθεση 7, το σημείο 7 δηλαδή, διότι έχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις αλλού οι ενδιαφερόμενοι. Πάω σε πάρουν αντιρρήσεις όχι. Και μερικές πληροφορίες τώρα. Ορισμοί που αποφάσισαν οι συντονιστές και συντονίστριες. Δεν θα γνωμοδοτήσουμε για το θέμα της ΙΤΡΑ και επιστημονικής συνεργασίας με την Ελιβετία στα πλαίσια του ορίζοντος 2020. Θα γνωμοδοτήσουμε όμως για την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής ΕΛΕΦ για την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη σφαιρικότερης αντιμετώπισης της έρωσης για τις μεταναστευτικές ροές. Ο Ζεράρντε Πρέιν, ο, ο συντάκτης της γνωμοδότησης. Για τον προπολογισμό του 16 οι συντονιστές συμφώνησαν το χρονοδιάγραμμα, το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα που δέχτηκε ο τριμερής διάλογος της 30 Μαρτίου και που θα το συζητήσουμε στο 11. Η Επιτροπή μας θα γράψει έκθεση για την εντολή του τριμερούς διαλόγου εν ώψη της Ολομελίας του Ιουλίου αμέσως μετά την παρουσίαση του προϋπολογισμού, την υποβολή του προϋπολογισμού από την Κομισιόν. Η έκθεση πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Οι συντονιστές συμφώνησαν για την πρόταση τροποποιητικού κανονισμού για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων μέσα στα πλαίσια του Πολδίπ. Είναι μια επιτάχυνση δηλαδή εδώ το 1% προχρηματοδότησης γίνεται 30% και αν αυτό γίνει με την απαραίτητη δυναμική μπορεί αυτό να καταλήξει σε ανεπάρκεια κανδυλίων μέχρι το τέλος του 2015. Επίσης συμφώνησαν να γίνει μια συλλογική απόσυρση των τροπολογιών για την αναθεώρηση, δηλαδή ψήφιση χωρίς τροπολογίες, ώστε να μην γίνει τριμερής διάλογος και απόρρια χρόνου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέξουμε ορισμένα πράγματα γιατί ως εισηγητής που δέχεται την απόσυρση των τροπολογιών ξέρω ότι όπου υπάρχει μεγάλη ανεργία η δυνατότητα απασχόλησης νέων είναι μικρή και γι' αυτό ό,τι ποσά και να διαθέσουμε. Και γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την κινητικότητα των νέων, να πάνε αλλού, να βρουν δουλειά αλλού. Επίσης έχουμε δύο αποστολάς, η μία στη Σικελία με 12 μέλη, 22, 23 και 24 Ιουλίου, σε συνεργασία με την Επιτροπή ΕΛΕΦ και για να προετοιμαστεί αυτή η αποστολή ο διευθυντής του Frontex θα κληθεί να κάνει μαζί μας μια ανταλλαγή απόψεων και επειδή ο κύριος Δεπρέ είναι εισηγητής της συντάξη της γνωμοδότησης για... θα μας πει και αυτός ό,τι ξέρει για τα λαμβανόμενα μέτρα ελέγχου των μεταναστευτικών ροών έτσι ώστε να υπάρχει εγγύηση του ασύλου, του δικαιώματος του ασύλου κλπ. Και δεύτερη αποστολή στην Εσθονία, 12 μελή και αυτή, στη Ρήγα 18 και 19 Ιουνίου. Τέλος, η επόμενη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών ΠροΥΠ και της Επιτροπής Ασφαλείας και Άμυνας στη αίθουσα Γιάνν 2Q2 ως προσθήκη στις τακτικές συνεδριάσεις του Επιτροπής ΠροΥΠ διότι προσέξτε το θα ψηφιστεί η κοινή έκθεση για τη χρηματοδότηση της πολιτικής κοινής άμυνας και ασφάλειας από την υποεπιτροπή εκείνη της ΕΠΕΞ και άρα αν θέλετε να υποστηρίξετε την εξαιρετική έκθεση θα σας παρακαλώ να προσέλθετε στις 14 Απριλίου 9 με 9.30 θα γίνει η ψυχοφθορία αυτή Τα πρακτικά της στις 16 Μαρτίου τώρα, εάν δεν υπάρξουν ιδιαίτερες παρατηρήσεις και αντιρρήσεις, μπορούν να εγκριθούν και περνάμε στις ψηφοφορίες. Ξεκινάμε από την έκθεση παριθμών 7. Ευκαιρίες πράξη, πράσινης ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρά τροπολογία 8 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ε, ο εξηγητής υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 1, τροπολογία 9, υπέρ ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφορία πέρας εγκρίνεται 19 προς 14. Παράγραφος 2, τροπολογία 12. Υπέρ εισηγητής, υπέρ. Κατά. Ε. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι, ας ελέγξουμε. Ηλεκτρονικό, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρασε. Ισοψηφία. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ ο συγκητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 2α14. Υπέρ ο συγκητής. Υπέρ. Κατά θες, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχεται το ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 16. Προφορική τροπολογία του κ. Τόρβαλ. Με καλύτερη νομοθεσία και με μείωση, μείωση του διοικητικού άρθρου στους υπερασυγητές υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπερασυγητές υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική α για την παράγραφο 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Ένα υπέρ ο υπέρ. Κατά. Δεν είδα να σηκώνονται χέρια ούτε στην μια περίπτωση ούτε την άλλη. Τροπολογία 1. Ελεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες, πέρασε. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 2. Συναυλία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται α, β υπέρ εισηγητής, 3, τοπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, το γίνεται. Αιτιολογική σκέψη α, τοπολογία 4, υπέρ εισηγητής, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία β, α, υπέρ εισηγητής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία, σε, τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν. Για το σύνολο του κειμένου. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Υπέρ. Με συγχωρείτε, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 32 προς 1. Τώρα, τέσσερα. Έκθεση παριθμών τέσσερα. Εννοεί αυτό. Υπέρ της έγκρισης της έκθεσης αυτής. Πολιετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, έκθεση το ΜΑ. Για την έγκριση της έκθεσης, υπέρ. Ας περάσουμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται ομόφωνα. 5. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. εδώ γιατί πραγματικά ανακοινώθηκε η κλίση μιας επιχείρησης. 2α. Τροπολογία 1 υπέρ ο Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3α. 2. Υπέρ ο Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 3. Τροπολογία 3. Υπέρ εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Ναι, 4. Υπέρ εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 3 σε 5. Υπέρ εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6, τροπολογία 6, υπέρ εισηγητής υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 7, τροπολογία 7, υπέρ εισηγητής. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7α, τροπολογία 8, υπέρ εισηγητής υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 δίτα, 9 υπέρ εισηγητής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 σ 10 υπέρ εισηγητής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 δ τροπολογία 11 υπέρ εισηγητής υπέρ κατά εγκρίνεται 7ε12 ε, υπέρ εσωτερικής υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 7F τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται. 8α14 υπέρ υπερ τις υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για το σύνολο του κειμένου. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 31 προς 3. η δική μου έκθεση, πρωτοβουλία για την ε, απασχόληση των νέων. Αποσύρω τις απολογίες μου και μου λένε ότι και ο κύριος Ιτουργκάης αποσύρει και τις κοινώς τις δικές του. Κατά συνέπεια, υπάρχει η τροπολογία 4. Τροπολογία 4 του κυρίου Σβέρ αποσύρθηκε όπως έχετε και αυτή. Οπότε δεν ψηφίζουμε. Υπ' αυτές τις συνθήκες πρωτοβουλία για επιστολή Προ τον πρόεδρο της Επιτροπής επασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων με αφορμή την απόσταση των πολιτιών μου εντόπισα την ε, δυσκολία έλλειψη πιστώσεων στο τέλο του 2015 εάν ο μηχανισμό συνεχίσει να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί τώρα. Με τι τροπολογίε που είχα υποβάλει και που απέσυρα ήθελα εδώ να επισημάνω και να επιστήσω την προσοχή στο ότι υπάρχει πρόβλημα την απασχόληση των νέων σε περιοχέ που είναι πολύ ψηλή δεν υπάρχουν θέσει εργασία. Και αν δεν υπάρχουν θέσει εργασία, πρέπει να ενθαρρύνουμε του νέου, μάλλον να πάνε εκεί που υπάρχουν δουλειέ. Για να ζήσουν την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία. Οι πολιτικοί ηθήνοντε πρέπει να λάβουν δράση εκεί που δεν υπάρχουν δουλειέ, να φροντίσουν να υλοποιηθούν οι απαραίτητε μεταρρυθμίσει για να πάρει μια ανάσα οικονομία όπω χρειάζεται και η ανταγωνιστικότητα να αναπτυχθεί και να δημιουργηθούν θέσει εργασία. Θα περάσουμε τώρα. Το σχέδιο επιστολής τώρα που θα ήθελα να αποστείλω στον πρόεδρο της Κομισιόν της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Έχετε κάποιες ε, παρατηρήσεις για το περιεχόμενο του. Πιστεύετε ότι μπορώ να το αποστείλω όσο έχει. Με την υπογραφή του πρόεδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του εισηγητή δεν έχετε αντιρρήσεις. Ωραία. Λοιπόν, θα αποσταλεί αυτή η επιστολή με τις ενθαρρυντικές σας ε, γνώμες, απόψεις και την υποστήριξή σας. Η κυρία Γουαρδία Σαμπάλ για τον προϋπολογισμό 2015, ε, ε, παρακαλώ. Δεν θα υπάρξει έκθεση, λέει ο πρόεδρος. Υπάρχει η επιστολή απλώς. Και η επιστολή καλύπτει και το περιεχόμενο της έκθεσης. Προσπαθώ λοιπόν σε αυτή την επιστολή να στείλω το μήνυμα της Επιτροπής μας. Κυρία Γουάρδια Σαβάλ, για την έκθεση στο σημείο υπαριθμών 8. Έχετε το λόγο. Αυτή η μεταφορά έχει να κάνει με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, κάτι το οποίο αναφέραμε ήδη προηγουμένως. Έχει ζητηθεί ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν η μεταφορά. Η κυρία Όλμαερ για το σημείο 9 άλλα τμήματα του προϋπολογισμού. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν μικρές ε, μεταφορές οι οποίες δεν έχουν προβληματικό χαρακτήρα προς την ε, αφορούν την Επιτροπή των Περιφερειών για την ενίσχυση της γραμματείας των πολιτικών ομάδων και στα πλαίσια της συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που περατώνονται σιγά σιγά και έχουμε περάσει σε αυτή τη μεταφορά πληστώσεων για να χρηματοδοτηθούν οι τρεις θέσεις στην ομάδα των φιλελευθέρων στην Επιτροπή των Περιφερειών. Αυτό δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και η δεύτερη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων αφορά την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Πρόκειται για μια μεταφορά δαπανών στον τομέα των επίπλων για μια ε, καταβολή κόστους μεταφοράς, ε, μετακόμισης, συγγνώμη. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο πρόβλημα το οποίο προξενείται από αυτές τις ε, μεταφορές πιστώσεων. Λοιπόν, ψηφίζουμε την πρώτη έκθεση για την Επιτροπή των Περιφερειών. Άρχεται η ψηφοφορία. Η πρώτη μεταφορά πιστώσεων. Ψήφισατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Η έκθεση για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, πάλι με ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται, 32-2. Κτηριακή πολιτική, ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κυρία Χολμάιερ, σε συμφωνία και με τους σκιώδεις εισηγητές επίσης, να σας πω τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχει δύο πύργους ήδη το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τώρα θέλει να έχει και ένα τρίτο πύργο για την στέγαση του προσωπικού του που βρίσκεται εκτός του κεντρικού κτηρίου αυτή τη στιγμή να μπορέσει να έρθει σε ένα χώρο που να είναι πιο κοντά αυτή τη στιγμή η υπηρεσία μετάφραση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου βρίσκεται σε ένα νοικιασμένο κτίριο και ο στόχος είναι να μπορέσει να υπάρξει ένα νέο κτίριο το οποίο θα μπορέσει να καλύψει 900 γραφεία. Αυτό θα καλύψει τις ανάγκες του προσωπικού προβλέπεται μέχρι το 2020. Μετά ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξει και μια νέα αντιμετώπιση. Ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα αυξήσει τον αριθμό των δικαστών και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη και πρόσθετου προσωπικού που θα συνοδεύσει αυτούς τους ε, δικαστές. Όλα αυτά λοιπόν έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί και με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η αύξηση της έκτασης κατά 30.000 τετραγωνικά μέτρα είναι αυτό το οποίο προβλέπεται. Αυτό το σχέδιο το είχαμε συζητήσει ήδη από το 2011 και γενικά η θέση που είχαμε πάρει ήταν θετική για το θέμα αυτό, ώστε να δώσουμε στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να πάρει τις 200.000 ε, ευρώ τα οποία ήταν απαραίτητα για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστος. Το κόστος λοιπόν τελικά θα είναι 131.800.000 ευρώ και θα έχουμε και την επιστροφή του κόστους χρηματοδότησης και επομένως με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα και σε σχέση με το κόστος θα μειωθεί και η ετήσια ε, επιβάρυνση κατά 6 εκατομμύρια μέσα σε 10 χρόνια με το γεγονός ότι δεν θα χρειάζεται να νοικιάζει πλέον κτίριο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και επομένως αυτό δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το ίδιο το Λουξεμβούργο, η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να δώσει όσο να τον καλύτερες συνθήκες για τα Ευρωπαϊκά Ένωση. Πήρε το οικόπεδο που θα χτιστεί ο νέος πύργος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ένα συμβολικό ευρώ. Αυτό φυσικά είναι πολύ θετικό. Αν γινόταν και κάτι τέτοιο στις Βρυξέλλες, με μεγάλη χαρά θα το δεχόμασταν. το Λουξεμβούργο αναλαμβάνει να είναι και, κτίριος, και κύριος του έργου το οποίο θα κατασκευαστεί. Προβλέπεται το 2019 να είναι έτοιμο το νέο κτίριο και το Λουξεμβούργο θα συμμετάσχει ιδιαίτερα στην διαδικασία κατασκευής του κτίριου και θα, θα εγγυηθεί την χρηματοδότηση του κτίριου αυτού και όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία θα επαναφέρει θα δώσει το κτίριο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Προβλέπεται μέχρι το 2036 να έχει αποπληρωθεί το κτίριο αυτό από το, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έτσι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραμένει στα πλαίσια της συμφωνίας που είχαμε συνάψει στο παρελθόν και δεν έχει αλλάξει τίποτα, παραμένει μέσα στα σωστά πλαίσια η όλη διαδικασία χρηματοδότηση. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω τώρα ως εισηγητής για τον προϋπολογισμό 16 των υπολείπων οργάνων. Δεν αμφισβητώ κανένα από τα στοιχεία που ανέφερε η κυρία Χολμάγερ, αλλά έχω ένα ερώτημα για τον προϋπολογισμό 17. η έγκριση που θα δώσουμε τι επιπτώσεις θα έχει στον προπολογισμό του 16. Διαβάζω στη σελίδα 8 του κειμένου που μας δώσανε. Το ποσό της αποζημίωσης για το ενίκιο που θα δοθεί στο λουξεμβουργικό κράτος θα είναι 22 εκατομμύρια το χρόνο μεταξύ 17 και 26 στην επόμενη παράγραφο λέει έχοντας υπόψη είναι το δημοσιονομικό άκτος που πρέπει να πληρώσει ακόμη το δικαστήριο από το 17 για τέτοια κτίρια, η συμπληρωμα... το συμπληρωματικό βάρος των προπλογισμών θα περιοριστεί σε ετήσιο ύψος 6 εκατομμυρίων ευρώ. Αν τα ερμηνεύω λοιπόν σωστά, δεν υπάρχει κόστος για το 16 στον προϋπολογισμό. Εκτός αν δεν καταλαβαίνω καλά μόνο από το 17 και μετά θα αρχίσουν να πληρώνουν ή μόνο το συμπλήρωμα του ενοικίου θα αρχίσει να πληρώνεται από το 17. Θέλω να το ξέρω και για το 16 για να ξέρω τι θα γράψω. Κύριε Εγώ βλέπω αυτά τα οποία έχω στα χέρια μου δεν θα υπάρχει πρόσθετο κόστος για το 2016. Από το 2017 θα ξεκινήσει και θα εγγραφεί στη συνεχεία στον προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία ελέγχθη. Νομίζω ότι το ίδιο το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να επιβεβαιώσει αυτά τα οποία αναφέρατε. Κύριε Ντεπρέ. Εντάξει, εγώ έχω εμπιστοσύνη στην κυρία Ολμάγερ, αλλά θέλω τη βεβαιότητα. Μήπως κανένας εκπρόσωπος του δικαστηρίου είναι εδώ. Να είμαστε συγκεκριμένοι. Έχουμε εδώ εκπρόσωπο του δικαστηρίου. Α, ε, να μας το πει εδώ πίσημα για να ξέρουμε όλοι τι επιπτώσεις θα έχουν όλα αυτά στον προπολογισμό του 16. Για το 17 είπαμε 22 εκατομμύρια το χρόνο περίπου 20% του προϋπολογισμού του κενοβουλίου. Βέβαια δεν έχει τιμή η δικαιοσύνη, έχει όμως κόστος. Ορίστε κύριε εκπρόσωπε του δικαστηρίου. Ναι, είμαι Γενικός Διευθυντής στο δικαστήριο, ευχαριστώ. θα ήθελα να καθησυχάσω τον κύριο Ντεπρέτα. Τα 22 εκατομμύρια που λέτε είναι η απόσβεση κτηρίων που έχει αναλάβει και χτίσει το δικαστήριο προηγουμένως. προηγουμένως. Αυτά τα 22 εκατομμύρια το χρόνο δηλαδή είναι οι προεκτάσεις που κάναμε στο παρελθόν επί του παλαιού κτηρίου. Ο τρίτος γύρος έχει μηδέν επίπτωση. Ο τρίτος, πύργος μάλλον, πύργος όχι γύρος, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Όταν χτιστεί τότε θα αρχίσει η αποπληρωμή και η απόσβεση. Και θα δείτε ότι από το 19-20 και όσο κρατήσει το δάνειο θα κρατάει και η απόσβεση. Δεν έχουν λοιπόν όλα αυτά επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του 16 κύριε εισηγητά μου. Τώρα το ερώτημά σας για τα 6 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια. Αυτό το είχαμε υπολογίσει τότε, το 11 δηλαδή. Για να δούμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ συνέχισης του ενοικίου, αν δεν χτίζαμε, από τη μία και χτισήματος του τρίτου πύργου. Αν οικοδομηθεί ο τρίτος πύργος τότε α, κατέτος 6 εκατομμύρια παραπάνω από ότι αν νοικιάζαμε το κτίριο στο Λουξεμβούργο. Μετά από 10 χρόνια αποσβαίνονται, αποσβέν, αποσβαίνεται και δεν θα έχουμε πια από τότε να πληρώνουμε ούτε τη διαφορά αυτήν. Τα στοιχεία που σας δώσαμε το 11 υπολογίζονταν με βάση τα δάνεια που θα κάναμε το 11 και όλοι μας οι υπολογισμοί βασίζονταν σε ένα δάνειο με επιτόκιο 5%. Γιατί θα θυμάστε ότι τα φτηνά δάνεια τότε είχαν τέτοιο επιτόκιο. Σήμερα νομίζουμε ότι επειδή βλέπουμε ακριβώς τι δαπάνες είχαμε, ότι μπορούμε να δανειστούμε με κάτω από 2% μεταξύ 1,5% και 2%. Και αυτό θα κάνουμε για τον τρίτο πύργο. Η διαφορά λοιπόν δεν θα είναι πλέον 6 εκατομμυρίων αφού δεν άλλαξε το ενίκιο. Η απόσβεση δεν θα είναι τόσο σημαντική γιατί θα είναι χαμηλότερο το επιτόκιο και η διαφορά θα είναι σχεδόν μηχανική και όταν αποσβεστεί, αν αποσβεστεί σε 15 χρόνια τότε δεν θα υπάρχει καμία διαφορά, δεν θα κοστίζει παραπάνω. Συμφέρει λοιπόν να χτίσουμε τον πύργο παρά να συνεχίσουμε το ενίκιο. Ευχαριστώ. Μα ποιος δανείζεται εδώ πέρα. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος. Με συγχωρείτε. Θέλω να απαντηθεί πρώτα η προηγούμενη ερώτηση που έθεσα. Θέσατε ένα ερώτημα κύριε Πρόεδρε. Ποιος δανείζει. Περιμένω την απάντηση. Ποιος δανείζεται μάλλον. Ποιος δανείζεται. Η Ένωση ισχύουν τα ίδια με αυτά που ίσχυσαν για τις προεκτάσεις του προηγούμενου κτηρίου. Επεκτάσεις που είχαν εγκριθεί από ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και εγκριθεί ως καλό πρότυπο το κράτος του Λουξεμβούργου μέσω μιας ειδική εταιρεία πηγαίνει στις αγορές και δανείζεται και εκείνο αποπληρώνει και το δικαστήριο πληρώνει το λουξεμβουργικό κράτος. Έτσι τα κάναμε όλα, με μηδενικό περιθώριο χωρίς καμία αποζημίωση λόγω των καλών μας σχέσεων με τις λουξεμβουργικές αρχές. Συν το οικόπεδο που δίνεται δωρεάν. Φτάνουμε στα όρια του παραλόγου βεβαίως, γιατί περνάμε από τεχνάσματα για να σώσουμε τις, ε, τα προσχήματα. Ξεχάστε αυτό το σχόλιο. Ο κύριος Ντεπρέ. Κύριε Πρόεδρε, να μην το ξεχάσουμε, γιατί τον ίδιο μηχανισμό θα τον απαντήσουμε και στην χρηματοδότηση του κτηρίου ΚΑΝΤ στο Λουξεμβούργο. Θα μας τα πει πολύ γρήγορα ο Γενικός Γραμματέας. Αν κατάλαβα καλά λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας δημοσιονομικός αντίκτυπος για το έτος 2016. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος ξεκινά από το 2017. Πρόκειται για μια σύμβαση ε, μίσθωσης ε, και πώλησης. Καλή συναλλαγή είναι, διότι το δικαστήριο θα είναι ιδιοκτήτης μια δεκαετία μετά την κατασκευή του κτηρίου θα έχει πληρώσει μόνο 6 εκατομμύρια επιπλέον ετησίω, διορθώστε με αν κάνω λάθο, και το συνολικό κόστο του κτηρίου θα είναι 10 επί 6, 60 εκατομμύρια, συν ε, την αποπληρωμή των επιτοκίων. Σωστά τα είπα. Από πλευρά προπολογισμού, ναι, όχι από το κόστο του κτηρίου. Το κόστο του κτηρίου θα είναι μόνον το κόστο κατασκευή, συν η τόκη. Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση, Πρόεδρε. Όπως είπαμε, το δημόσιο χρέος του μεγάλου δουκάτου του Λουξεμβούργου θα αυξηθεί από αυτή την επένδυση, γιατί πρόκειται μια επένδυση του Λουξεμβουργιανού κράτους. Δεν ξέρω από άποψη Μάστερ τι μπορεί να δώσει, αλλά από την πλευρά των δημοσιονομικών του κράτους μάλλον εξωτερώνεται Κοιτάξτε, όταν είχαμε κάνει την πρώτη μας προέκταση είχαμε ένα πρόγραμμα 400 ε, εκατομμυρίων ευρώ, αλλά το Λεξουμβουργιανό κράτος δεν τα ήθελε αυτά στον ε, προπολογισμό του. Γι' αυτό δημιουργήσε μια ιδιωτική εταιρεία, ε, μεσητική, και ε, τα περνάει από εκεί. Όχι, όχι, μηδενικό περιθώριο για τις αρχές του Λουξεμβούργου. Κοιτάξτε, πρόεδρος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα ήταν ίσως πιο απλό πράξεις μας να συνάδουν και με την πραγματικότητα. Περνάμε από απίστευτα τεχνάσματα και πρέπει να τα εξηγήσουμε μετά αυτά στους συμπολίτε μας. Πρέπει να έχει κανείς την τόλμη. Αλλά λογικό είναι να προκαλούμε και υποψίες σε κάποιες περιπτώσεις. Εφόσον πρόκειται για το δικαστήριο βεβαίως, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κύριε Δενανό, Πρόεδρε από χρόνια η Ευρώπη έπρεπε να έχει την ικανότητα να εφευρίσκει. Ε, τώρα έχουμε τέτοιες καταστάσεις παραλόγου, ας τα σκεφτούμε καλύτερα για το μέλλον. Ναι, να δανειζόμαστε αλλά με σύνεση. Για να επενδύουμε και όχι για να χρηματοδοτούμε δαπάνες λειτουργίας. Συμφωνούμε απολύτως, αν πρόκειται περί αυτού. Εγώ μαζί σας. Κυρία Χολμάγερ, να ψηφίσουμε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία έρχεται. Έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 27 ψηφί υπέρ, 2 κατά. Περνάμε τώρα στον προϋπολογισμό του 2016 που είναι ακόμα εν προετοιμασία και θέλω να σας κάνω και μια, ένα απολογισμό του τριγωνικού διαλόγου στον οποίο συμμετέσχα μαζί με την κυρία Γουάρδια Σαβάλ η οποία ενισχύεται για το 2015 και τον κύριο Φερνάντες για το 2016 και τον κύριο Ντεπρέ για τα άλλα τμήματα του 2016. Καταρχήν για την κατάσταση των πληρωμών πήραμε μια δήλωση σε σχέση με την κατάσταση των πληρωμών και υποχρεώσεων για το 2014. Έχουμε 24 δισεκατομμύρια απλήρωτους λογαριασμούς παρά τα 4 και κάτι δισεκατομμύρια που επιτύχαμε σε, στον τριγωνικό διάλογο στο τέλος του 2014. Αναφέραμε στην ε, Κομισιόν ότι περιμένουμε πάντα το σχέδιο για την εξόφληση όλων αυτών των λογαριασμών που εκκρεμούν. Αυτή ήταν μια δέσμευση που είχε αναλυφθεί στο τέλος του 2014 μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Αναμένουμε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα για την αποπληρωμή όλων αυτών των υποχρεώσεων και περιμένουμε να δούμε και μία συζήτηση σε σχέση με το αποδεκτό επίπεδο που θα πρέπει να έχουν αυτές οι απλή, αυτοί οι απλήρωτοι λογαριασμοί. Συμφωνήσαμε λοιπόν να υπάρξει μια παρουσίαση ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμών του συνοπτικού πίνακα για τις πληρωμές. Αυτό θα λάβει χώρα στις 16 Απριλίου, τις 9.30 με 10.30 το πρωί. Και η κυρία Γεώργεβα η αρμόδια αντιπρόεδρος για τα θέματα του προϋπολογισμού θα είναι παρούσα σε αυτή την παρουσίαση. Επίσης, καταλήξαμε με θετικό τρόπο σε σχέση με μια συνεδρίαση της διαθεσμικής ομάδας πριν από το τέλος Μαΐου, ώστε να συζητηθεί το σχέδιο αυτό εκαθάρισης των ε, απλήρωτων λογαριασμών. Μέχρι τότε μπορούμε να συνεχίσουμε τις άτυπες επαφές για να εξασφαλίσουμε ότι το έγγραφο αυτό είναι πράγμα αυτό το οποίο περιμένουμε και απλό και δεν θολώνει περισσότερο τα νερά και στη συνέχεια μετά από αυτήν την ομάδα υψηλού επίπεδου θα ακολουθήσει ίσως ένα τριγωνικό διάλογο για να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα για την αποκληρωμή των λογαριασμών αυτών που εκκρεμούν. Επίσης θα έχουμε και μια ανταλλαγή απόψε για τις κατευθυντήρες γραμμές του 2016 είχαμε μάλλον αυτή τη συζήτηση, η οποία ήταν επικοδομητική, το Συμβούλιο δείχνει να εμφορείται από καλές προθέσεις. Θα δούμε βέβαια ποια είναι η πραγματικότητα όταν το Συμβούλιο εκφράσει την άποψή του σε σχέση με το προσχέδιο που θα μας υποβάλει η Κομισιόν στις αρχές του έτους, του καλοκαιριού. Έχουμε επίσης δει και το χρονοδιάγραμμα των ε, συνδιαλλαγών. Θυμόμαστε όλοι πώς πήγαν οι συνδιαλλαγές του 2014. Ελπίζουμε ότι θα είναι σε υψηλότερο επίπεδο η εκπροσώπηση του Συμβουλίου στην τρέχουσα συνδιαλλαγή. Αλλιώς θα στείλουμε και εμείς τους συνεργάτες μας και όχι οι βουλευτές. Το Συμβούλιο τόνισε τη θέλησή του να τελειώσει αυτή η διαδικασία <clears throat> στις 13 Νοεμβρίου. <clears throat> Αυτό είναι μια ημερομηνία η οποία είναι γουρλίδικη, αλλά Η τελευταία ημερομηνία θα είναι η 18, 18 Νοεμβρίου. Το Συμβούλιο, επειδή θα έχει μεγάλο φόρτο εργασίας, ήθελε να τελειώσει στις 13 του Νοεμβρίου. Εμείς είπαμε ότι αν θέλετε να το κάνετε αυτό θα πρέπει να δεχτείτε τη θέση του Κοινοβουλίου, αλλιώς θα πρέπει να συνεχίσετε τη συνδιαλλαγή μέχρι τις 18 που είναι η καταληκτική ημερομηνία, ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί ένας περαιτέρω τριγωνικός διάλογος αν αποτύχει αυτό το εγχείρημα. Αναφερθήκαμε <clears throat> επίσης στους διορθωτικούς προϋπολογισμούς 1 και 2, μας είπε η κυρία Γουάρδια Σαβάλ ότι για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Στρατηγικών Επενδύσεων θα πρέπει να περιμένουμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να δούμε τι θα προκύψει και τότε ο διορθωτικός προϋπολογισμός θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη. Για το δεύτερο διορθωτικό προϋπολογισμό έχουμε την έκθεση Όλμπριχτ και Τομά. Λογικά θα ψηφίσουμε στα τέλη Απριλίου για, τον... για τη διορθώση αυτή και έχουμε επίσης μια ανταλλαγή απόψεων για την μείωση κατά 5% των θέσεων στο οργανόγραμμα των ευρωπαϊκών οργάνων, όπου αναφέρθηκε ότι είναι καλό το να μειωθούν κατά 5%. Αλλά αν το αποτέλεσμα είναι η εξωτερική ευσιοσμένη υπηρεσιών, αυτό δεν έχει κανένα απολύτως θετικό αποτέλεσμα. Αν το κάνουμε μονάχα για να ευχαριστήσουμε την κοινή γνώμη, αλλά τελικά πληρώνουμε ε, για παροχή υπηρεσιών στα θεσμικά όργανα που γίνεται για να αντικατασταθούν οι θέσεις εργασίας που χάνονται, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι σαν μια επιχείρηση που κάνει μια επένδυση στη θέση της επένδυσης που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς οι και μετά πρέπει να πληρώνουμε νίκια αντί να κάνουμε επένδυση σε ένα κτίριο. Λοιπόν, επιστήσαμε την προσοχή της Κομισιόν <clears throat> στο σημείο αυτό και του Συμβουλίου εναντίον των ε, δράσεων αυτών των ενεργειών που είναι απλώς δράσεις βιτρίνας και δεν έχουν κανένα πραγματικό αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν για τον τριγωνικό διάλογο τον... ο οποίος έγινε χθε. χωρίς μικρόφωνο. Έχετε κάποιες παρατήρησεις σχετικά? Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο σχετικά. Και ερχόμαστε τώρα στα πιλωτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τον προϋπολογισμό 15 και 16. Με εισηγήτρια την κυρία Γουάρδια Σαβάλ και τον κύριο Φερνάντες. Θα τους δώσω λοιπόν το λόγο. Κύριε Φερνάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Τα πιλωτικά προγράμματα είναι μια ευκαιρία να μπορέσουν οι βουλευτές με κάποιες προτάσεις για δράσεις να συμμετάσχουν και να προκαλέσουν τη δημιουργία σημαντικών προγραμμάτων. Τα πιλωτικά προγράμματα έχουν ένα περιορισμένο περιθώριο αλλά έχουμε εδώ ένα δικαίωμα πρωτοβουλίας και μπορούμε να προχωρήσουμε με προγράμματα που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητές μας. Μία από αυτές είναι ο στόχος της απασχόλησης. Έχουμε χιλιάδες α, θέσεις απασχόλησης που πρέπει να καλυφθούν στην Ευρώπη διαρκώς και υπάρχουν διάφορα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις εδώ για την απασχόληση των νέων, αλλά δεν υπάρχει κανένα πιλωτικό πρόγραμμα για αυτούς των άνω των 30. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ευκαιρία και ήθελα να εκφράσω αυτήν την ε, πρόθεση σε σχέση με τα πιλωτικά προγράμματα τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις μπορεί να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα χειροπιαστά βήματα. Έχουμε ένα έγγραφο που καταγράφει την κατάσταση των πιλωτικών προγραμμάτων που ήδη τρέχουν. Ένα έγγραφο εργασίας που χρησιμεύει ως διευκρίνηση ε, για οποιαδήποτε πορεία είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Καρτία Όχι, ο Ζούμπιχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα ερώτημα για τον προπολογισμό του 2016. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ενεργείας στην Ευρώπη και η Επιτροπή μας είχε προ... προτείνει να υποστηρίξουμε ένα πρόγραμμα για τις ε, γυναίκες οι οποίες θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν για τη δημιουργία ε, επιχειρήσεων. Αυτό είναι πολύ καλό αν οι γυναίκες μπορούν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις όπου ιδιαίτερα στις χώρες όπου υπάρχει μεγάλη ανεργία. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα έχει θετικό χαρακτήρα. Περιμένω τώρα από την Κομισιόν να μας πει τι γίνεται με το πρόγραμμα αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει και στο οποίο δώσει τη συνένεσή του και το α, Συμβούλιο ε, μαθαίνω όμως ότι η κυρία Μπιενκόφσκα έχει αποστασιοποιηθεί από αυτό το πρόγραμμα. Εμείς θα θέλαμε όμως να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τη στάση της Κομισιόν σε σχέση με αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι είναι μια πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο για να αντιμετωπιστεί η ανεργία και δεν είναι κάτι το οποίο η Κομισιόν μπορεί να το απορρίψει χωρίς καμία δικαιολογία και χωρίς να επιστήσει την προσοχή μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν αμφιβάλλω ότι θα σας υποστηρίξουν στην αίτησή σας αυτή. Κάποιος άλλος θέλει να λόγο για τα πιλωτικά. Συγγνώμη που σας ενοχλώ λιγάκι ως πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που ήθελαν να κάνουν, να υποβάλουν ένα πιλωτικό σχέδιο για την κινητικότητα των νέων προτείνοντας ότι οι νέοι ηλικίας 18 ετών να μπορούν να μεταβούν τουλάχιστον για ένα χρόνο σε μια χώρα που δεν είναι η δική τους χώρα για ένα συμβόλαιο μαθητείας. Και υποθέτω ότι στις χώρες όπου θα μεταβούν θα μπορέσουν να τις υποδεχτούν οι οργανισμοί εκπαίδευσης και κατάρτισης για να μπορέσουν να συμπληρώσουν την ε, εκπαίδευσή τους σε διάφορα θέματα που τους ενδιαφέρουν και επίσης να τους βοηθήσουν να μάθουν τη γλώσσα της χώρας όπου πηγαίνουν. Θα είναι λοιπόν συμβόλαιο μαθητείας τουλάχιστον ενός έτους με την απότερη ελπίδα ότι κάποια μέρα θα μπορέσει να υπάρξει σύγκληση της νομοθεσίας για τις μαθητείες ώστε να υπάρχει ενιαία νομοθεσία που να μπορεί να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα επανέλθω λοιπόν στο θέμα αυτό ή αυτό το πιλωτικό θέμα το οποίο προσπαθούμε να μορφοποιήσουμε. Γιατί πρέπει να ανταποκριθούμε στις αιτήσει των νέων. Όχι μόνο τον το να ξαναδίνουμε χρήματα στα κράτη-μέλη για να συνεχίσουν τις ενέργειές τους που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες αλλά έχουν περισσότερο χαρακτήρα προβολής προς τα έξω και δημοσίων σχέσεων και όχι πραγματικής κατάρτισης. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό το θέμα και θα με συγχωρήσετε αν είμαι επίμονος άμα το παρακάνω πέστε μου το. Άλλες αιτήσει για λήψη του λόγου. Όχι. Ερχόμαστε τώρα στο τμήμα 1 προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2016 και το λόγο έχει ο κύριος Ντεπρέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να θυμίσω ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε αποδεχτεί τις μεγάλες γραμμές των γράφων που είχα προτείνει και που χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι για τον ορισμό του ποσοστού αύξησης των δαπανών του Κοινοβουλίου για το 2016 δεχτήκαμε διαχωρισμό μεταξύ αυτού που ονομάζω με απλό τρόπο τα απλά έξοδα λειτουργίας και τα έκτακτα έξοδα επενδύσεων. Νομίζω ότι από αυτού υπήρξε γενική συμφωνία εντός της Επιτροπής μας. Τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά για το ποσοστό αύξησης των ε, τρεχών δαπανών, των τρεχόντων εξόδων. Είπαμε το ποσοστό αυτό να είναι στο ε, μέγιστο σε ανώτατο όριο 1,9%. Το αποφασίσαμε αυτό σε ανεπίσημη συνάντηση και με τους κοιόντες εισηγητές όλων των πολιτικών ομάδων και είπαμε ότι κατά τη συνδιαλλαγή με το Προεδρείο θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσει ξεκινώντας με ένα ποσοστό αύξηση για τον προπολογισμό για τις τρέχουσες δαπάνες 2016 1,3 1,3, κάτι που είχε προτείνει έτσι αλλιώς μια από τις πολιτικές ομάδες και κατά δεύτερον σε ό,τι αφορά το ε, ποσό των δαπανών λειτουργίας είπαμε να ασχοληθούμε κυρίως με τα θέματα της ασφάλειας των κτηρίων και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις με την αντιπροσωπεία που προεδρεύετε εσείς κύριε Πρόεδρε και τι προέκυψε από τις συναντήσεις μας ως τώρα σε αυτό το στάδιο καταλήγουμε ε, στο σχέδιο του προπολογισμού το φθινόπωρο έτσι κι αλλιώ, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε το γενικό πλαίσιο από τώρα, εντό του οποίου θα εντάξουμε τα κεφάλαια που πρέπει να γίνουν αυξήσεις και εκεί που θα πρέπει να γίνουν cuts, όπως λέμε στα αγγλικά, δηλαδή δημοσιονομικές περικοπές. Αυτό ήταν το γενικό πλαίσιο και απασχόλησε την πρώτη συνάντηση τη συγγελαγή. τώρα από την πλευρά τη αντιπροσωπεία του Προεδρείου. Σε ό,τι αφορά τι δαπάνε λειτουργία. Το ποσοστό αύξηση των δαπανών που ζητούν για το 2016 σε σχέση με το 2015 είναι 2,2%. Η δική μας αντιπροσωπεία ξεκίνησε από το 1,3% και κάποια στιγμή μετά από διάλογο πρότεινα να περιοριστούμε στο 1,6 κατανατατόριο. Δηλαδή να αυξήσουμε την δική μας πρόταση από το 1,3 στο 1,6 και αντιπροσωπεία του Προεδρείου να μειώσει τη δική της κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. Εμείς δηλαδή κάναμε το 1 τρίτο και εκείνη το 2 τρίτο της διαδρομής για να συναντηθούμε. Βεβαίως δεν συμφωνήσαμε στις ε, έκτακτες δαπάνες για τον προπολογισμό του 2016 και για την ασφάλεια των κτηρίων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αυτές θα περιοριστούν σε ένα ε, μέγιστο πόσο 15 εκατομμυρίων ευρώ. Και περιμένουμε πρωτού καθοριστεί ε, οριστικά το ποσό η έκθεση του Γενικού Γραμματέα που θα εξηγεί το σύνολο των δαπανών που θα προγραμματιστούν θα αιτιολογεί το κόστος. Εδώ έχουμε φτάσει στο επίπεδο συνδιαλλαγή με το Προεδρείο ο τριμερή διάλογο τώρα. Έλαβα τροπολογίε για το σχέδιο έκθεση. Θα τι εξετάσω. Θα τι εξετάσω με του σκιώδεις εισηγητέ. σε συνάντηση μεταξύ δύο και τρει σήμερα και μετά θα έχω και μια πρώτη συνάντηση με του κοιότητες εισηγητέ για την ε, οικονομική για τη φύση των οικονομιών, την, το χαρακτήρα των οικονομιών που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Ο Γενικό Γραμματέα θα παραστεί και στην επόμενη συνάντηση συνδιαλλαγή με μια πρόταση για μείωση 10 εκατομμυρίων ευρώ για τι ε, τρέχουσε δαπάνε και θα τα δω ε, ευθύ αμέσω στη συνάντηση με του συναδέλφου για να προστατεύσουμε τι προτεραιότητέ μα και τι οικονομίε επί του προπολογισμού μα. Το να φτάσουμε σε συμφωνία με το Προεδρείο σε μια συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, 23 ή 24. Και μετά να ψηφιστεί η έκθεση μου στην Ολομέλεια, στη Σύνοδο του τέλους Απριλίου. Αυτά μπορώ να πω σε αυτή τη φάση, Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Ντεπρέα, κύριος Μάγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτές τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι σε ό,τι αφορά τα θέματα της ε, της ε, δημιουργίας του προϋπολογισμού θα πρέπει να διατηρήσουμε τα όρια του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως ακριβώς τι γίνεται ώστε να μπορούμε να ε, αποφασίσουμε για τον προϋπολογισμό. Η τιμαριθμική αναπροσ... αναπροσαρμογή θα αφορούσε κανονικά 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό όμως δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Δεν θα χρησιμοποιηθεί, οπότε αυτό μας δίνει, συγγνώμη, δεν χρησιμοποιηθεί, αυτό μας δίνει ένα αποθεματικό το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να μην υπάρξει εξάντληση των προϋπολογισμών. Και επομένω, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η πρωτού κάνουμε αυτή την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού να σκεφτούμε καλύτερα για τις προτεραιότητες και τις ανάγκες που έχουμε. Αλλιώς καταλήγουμε σε ποσά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γι' αυτό η δική μας πολιτική ομάδα θέλει να κρατήσει τον προϋπολογισμό στα πλαίσια του πληθωρισμού και μόνο, το 1,3% που ισχύει. να κρατήσουμε στο 1,3%. Έχουμε λοιπόν και άλλα ποσά τα οποία οφείλονται. Αναφέρθηκα στα 12 εκατομμύρια ευρώ, αλλά 2 εκατομμύρια αφορούν τα άτομα ε, που φεύγουν από τις θέσεις απασχόλησής τους γιατί μειώνουμε το οργανόγραμμα κατά 5% αναφέρθηκε και η κυρία Όλμαερ σε αυτό. Βλέπουμε ότι είχαμε αποφασίσει το 2014 ένα αποθαματικό και δεν θα έπρεπε να συζητάμε μονάχα για τα μικρά ποσά. Και ένα περαιτέρω θέμα είναι το θέμα της συζήτησης με τον ερωτήσεων προς την Κομισιόν. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες ερωτήσεις. Αν, αν τα υπολογίσουμε όλα αυτά, κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ. Ξέρω άτομα τα οποία ήταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από 10 χρόνια και μέχρι τότε εκείνη την εποχή είχαμε 50 περίπου ερωτήσεις το χρόνο και τώρα έχουμε χίλιες ερωτήσεις. Αυτό λοιπόν είναι υπερβολικό το τεκμηριώνει και το Vote Watch. Νομίζω ότι και αυτό μας βλάπτει. Θα πρέπει να είμαστε πιο λογικοί και να μην αποδιόμαστε μονάχα σε δράσεις δημοσίων σχέσεων. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό για το οποίο έχουμε εκλεγεί και το οποίο είναι η νομοθετική μας εργασία. Μπορούμε να κάνουμε σημαντικές ε, εξοικονομήσεις για τις, για τις ε, ερωτήσεις προς την Κομισιόν καλύπτεται το 1% του προϋπολογισμού μας. Μπορούμε να το μειώσουμε αυτό το κονδύλι κατά 50% τουλάχιστον. Υπάρχουν και άλλα αποθεματικά τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε σημαντικές εξοικονομήσεις με τη μείωση της γραφειοκρατίας. Έχουμε λοιπόν σημαντικά αποθεματικά τα οποία μπορούμε να τα κινητοποιήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε υποφελώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μάγκα, κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντέπρε για τις ενέργειες που έχει κάνει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικά όλα αυτά. Μας ενδιαφέρει να επιτύχει και τα σωστά αποτελέσματα. Από την πλευρά του ΕΛΚ υπάρχει μια κόκκινη γραμμή την οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε. Αυτό είναι το 20% των συνολικών διοικητικών δαπανών. Αυτό είναι κάτι το απόλυτο μέγιστο που μπορούμε να έχουμε. Θέλουμε να έχουμε ε, εξοικονομήσεις ιδίως στον τομέα της ε, ασφάλειας. Νομίζω ότι με την εσωτερικοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγάλη εξοικονόμηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας να πάρουμε τα αντίστοιχα μέτρα το ταχύτερο δυνατό και να τα εφαρμόσουμε και είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα ασφαλείας κατεπηγόντως είναι κάτι το αποφασιστικό για όλους μας και φυσικά θα πρέπει να συζητήσουμε τις ε, πιθανές περικοπές με τον Γενικό Γραμματέα και επίσης θα πρέπει να δούμε ποιες εξοικονομήσεις είναι δυνατές στην πολιτική κτίριων με το να μειώσουμε τον νίκη που πληρώνουμε με την αγορά κτίριων. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο για ε, εξοικονόμηση και πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ότι βρίσκεται στο περιθώριο μας μέχρι το 20% για να αγοράσουμε τα κτίρια αυτά και επομένως να μειώσουμε το κόστος μίσθωσης. Υπάρχουν λοιπόν πολλαπλές δυνατότητες εξοικονόμησης στον τομέα αυτό και εγώ θα ήθελα να κάνουμε μια προσπάθεια να επιτύχουμε όσο το δυνατόν με περισσότερες μειώσεις λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση της ε, λιτότητας που ισχύει στα, σε πολλά από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω να ζητά άλλος κανείς το λόγο. Κύριε Ντεπρέ, ο Γκάγερ. Ευχαριστώ. Τρία ερωτήματα θέλω να θέσω στον κύριο Γκάιερ, καθώς τεχνικού χαρακτήρα. Κατάλαβα καλά ότι ο τελευταίος προϋπολογισμός μας είχε 71 εκατομμύρια πλεόνασμα. Επομένως έχουμε κάποιο περιθώριο στον προϋπολογισμό. Γιατί υπάρχει κάποιο κόστος το οποίο ούτως ή άλλως πρέπει να το αποπληρώσουμε. Αυτό είναι ένα πρώτο ερώτημα. Επίσης άκουσα τα επιχειρήματα του κυρίου Μάγκα για την, ε, ε, και για την ασφάλεια και τις άλλες εξοικονομίες. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε την μείωση του προσωπικού η οποία υποτίθεται θα μας φέρει εξοικονομήσεις. Υπάρχει αυτή η διαθεσμική συμφωνία για τα 5%. Οι πολιτικές ομάδες τονίζουν ότι αυτό δεν θα πρέπει να θίξει το προσωπικό των πολιτικών ομάδων. Και γι' αυτό μου φαίνεται απαραίτητο να κάνουμε τις απαραίτητες συζητήσεις για να προετοιμάσουμε τις αποφάσεις μας στον τομέα αυτό. Στην πρόταση τώρα του Γενικού Γραμματέα περιλαμβάνεται η μείωση λόγω της μείωσης του προσωπικού που απορρέει από την διαθεσμική απόφαση. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Έχετε κάνει μια πρόταση. Είπατε ότι υπάρχουν πάνω μια προσθήκη 15 εκατομμύρια για λειτουργικό κόστος. Μπορείτε να μου πείτε από πού ακριβώς προέρχονται αυτά τα 15 εκατομμύρια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Διότι στους Ελλάδους θα συναντηθούμε ισχυώδης και θα συζητήσουμε τις συμβαστικές προτάσεις για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά από πολιτικής σκοπιάς θέλω να πω, είναι σημαντικό για μένα, ε, να ακουστεί ότι πρέπει να περιορίσουμε τον προπολογισμό και να προσπαθήσουμε να ξαναδούμε τις δαπάνες μέσω των προβλεπόμενων μηχανισμών για την χρηστή διαχείριση του προπολογισμού και των ε, δημόσιων δαπανών. Οι Γερμανοί συνάδελφοι αυτή τη λιτότητα δεν τον εφαρμόζουν εντός του προπολογισμού του Κοινοβουλίου. Ε, το βρίσκω αρκετά ε, εντυπωσιακό αυτό, ενώ ισχύει η διαλυτότητα για τα κράτη του Νότου. Πρέπει λοιπόν να περιοριστούν οι διασπαθήσεις και να ε, γίνουν ε, οικονομίες. Ο αντιπρόεδρος Ασόλη έκανε προτάσεις για περικοπές και 10 εκατομμύρια οικονομίας που μας ε, υποσχέθηκαν. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ακόμη περισσότερα, διότι η κοινή γνώμη μας κοιτάζει με ιδιαίτερη προσοχή. Ο τρόπος που μπορεί να αυξάνουμε το κόστος της πολιτικής είναι σφάλμα που θα πληρώσουμε μετά όλοι. Αλλά έχουμε την δυνατότητα να λάβουμε κρίσιμες αποφάσεις. Ευχαριστώ. Δεν βρέπω άλλος να ζητά το λόγο. Η κυρία Χολμάγερ. Με συγχωρείτε. Για την τελευταία παρατήρηση είπα ότι αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθούσε το παράδειγμα του Ιταλικού Κοινοβουλίου θα είχε ο καθένας μας 10 ε, συνεργάτες. Βέβαια ακόμα περισσότερους έχουν στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Προφανώς έχουν πολύ περισσότερη εργασία από ό,τι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί λοιπόν συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται ιδιαίτερα έντονα. Αυτό δεν είναι μονάχα με τις ερωτήσεις προς την Κομισιόν όπως λέει το Vote Watch, το οποίο και εμένα με ενόχλησε. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί βουλευτές οι οποίοι εργάζονται ιδιαίτερα έντονα όταν έχουν παραδείγματο ένα δύσκολο θέμα να διεκπαιρεώσουν, όπω παραδείγματο χάρη Ζεραντεπλέ με τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πολύ σπάνια λαμβάνουν το λόγο, δεν παρουσιάζονται στις επιτροπές όπως η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε λίγο καλύτερα και για την παρουσία και την δραστηριότητα των βουλευτών. Και φοβάμαι ότι και εγώ πρέπει να αρχίσω να κάνω απεξηγήσεις ψήφου για να με γράφει το Vote Watch. Υπάρχει πράγματι η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε πρόσθετο φόρτο εργασία. Άμα δείτε ότι πρέπει εμεί να ελέγχουμε τι κατεξουσιοδότηση πράξη και άλλα θέματα, καταλαβαίνετε ότι οι βουλευτέ αλλά και οι γραμματείε των επιτροπών μα χρειάζονται επαρκέ προσωπικό και οι πολιτικέ ομάδε εξ, εξάλλου. Και δεν τρέπομαι να το πω αυτό καθόλου. Έχουμε κάνει πολλέ εξοικονομήσει σε ό,τι αφορά την διερμηνία. <clears throat> και πρέπει να λάβουμε υπόψη και το προσωπικό, όπως είπε το Συμβουλίο, το οποίο δεν βρίσκεται <clears throat> στο οργανάγραμμα. Εμείς έχουμε κάνει σημαντικές ε, εξοικονομήσεις και στα θέματα μετάφρασης. Ο κύριος ε, Γκαέρ επίσης έλαβε το λόγο προηγουμένως και είπε ότι αυτό το οποίο αφορά στις ε, πολιτικές ομάδες δεν πρέπει να υπολογίζεται μέσα στον προϋπολογισμό της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί δεν μπορεί κανείς να υποβάλει την πολιτική εργασία των βουλευτών στις, στους περιορισμούς του διοικητικού κόστους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξω αυτά που λέει ο κ. Γκάιερ, ότι στον προϋπολογισμό το κόστος το οποίο πρέπει να μειωθεί θα πρέπει να αφήσει απ' έξω το πολιτικό προσωπικό, το προσωπικό των πολιτικών ομάδων. Αυτό είναι πολιτικό προσωπικό δεν είναι τμήμα της γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να το επαναλάβω λοιπόν ότι αυτό το έχει δεχτεί η Κομισιόν στο παρελθόν, δεν πρέπει να το λησμονήσει. Είναι καλό να το έχουμε υπόψη μας για τον επόμενο χρόνο. Μάλιστα. Σας υπενθυμίζω ότι εχθές από το σεμινάριο καταλήξαμε ότι υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης των αποδοτικότητας. Και μεταξύ των μελετών που μπορεί να ζητήσει η Κομισιόν ή η Επιτροπή μας θα έπρεπε να γίνει μία αποτίμηση ακριβώς και αποδοτικότητας. Και φαίνεται ότι τα κριτήρια αξιολόγησης της αποδοτικότητας μπορούν να καταλήξουν σε αρνητικά συμπεράσματα και σε επιπτώσεις σε καταχρήσεις. Και άρα πρέπει να τα ξαναδούμε ορισμένα από αυτά. γιατί μερικά από αυτά είναι άχρηστα. Τέλος πάντων, κύριος Χριστοφόρου. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο, αλλά πιστεύω ότι έχω μια διαφορετική προσέγγιση. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Ευρώπη κρίνεται από τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ευρώπη κρίνεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αποδοτικότητα τη και από την τελεσματικότητα τη στο σύνολο. Και δεν πιστεύω κανένα Ευρωπαϊο πολίτη και κανένα λαό να ασχολείται αυτή τη στιγμή εάν θα περικόψουμε ή αν θα δώσουμε 2,2% αύξηση στον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 1,9%. Αυτό που για μένα έχει σημασία είναι να μην γίνονται δαπάνε για χάρη των δαπανών και εμεί να μην κάνουμε περικοπέ για χάρη των περικοπών. Εάν πράγματι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ανάγκη για αύξηση 2,2% να το κρίνουμε στο έργο του. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν κάνεις περικοπές στο τέλος και να μην αποδώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η γραμματεία θα έρθουν να μας πούνε ότι είναι απότοκο γιατί τους περικόψαμε και τους περιορίσαμε τις δυνατότητες. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι να δώσουμε τα όπλα και τα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αποδώσει πιθανές μειώσεις τελικά να αποβούν σε βάρος του ελέγχου, σε βάρος της αποδοτικότητας, σε βάρος της αποτελεσματικότητας που αυτό θα κρίνει ο πολίτης. Πιστέψτε με, κανένας Ευρωπαίος πολίτης δεν παρακολουθεί σήμερα εάν ο προπολογισμό πήγαινε 2,2% επάνω ή 1,9%. Και να σα πω και κάτι, και 100% να κόψουμε τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα πάρουμε πίστοση από του πολίτε. Θα μα πούν οι πολίτε ότι για να το μειώνετε στο μηδέν σημαίνει ότι κάνατε καταχρήσει τα προηγούμενα χρόνια και δεν το μειώνατε από τα προηγούμενα χρόνια. Άρα μας ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, το αποτέλεσμα και το έργο που θα παραχθεί και πιστεύω ότι δεν πρέπει να κάνουμε ανατολίτικο παζάρι για 0,5 ή 0,8 για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, νομένου ότι πιστήκαμε ότι θα αποδώσει αυτός ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Cela est juste certainement, mais comment Το θέμα είναι βέβαια πως μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερα λεφτά. Κύριο Στάραντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις και ένα παράδειγμα. Όπως είπα πολλές φορές, εμείς υποστηρίζουμε ως ομάδα την σόφρονα αντιμετώπιση του εισηγητή στα δύσκολα προβλήματα του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμφωνούμε απόλυτα με την ανάγκη να παρακολουθούμε πολύ καλά τις προτεραιότητες και τις ε, πολιετές τις ε, και των προηγούμενων κοινοβουλίων. Πρέπει να πληροφορήσω την Επιτροπή μας ότι οι πράσινοι είναι κατά της αύξησης για τις αμοιβέ των ε, συνεργατών των βουλευτών, παρά το γεγονός ότι εγώ προσωπικά έχω αντίθετη άποψη με την ομάδα μας και η ομάδα μας αντιμετωπίζει με πολύ σκεπτικισμό τις αυξήσεις στον προϋπολογισμό της πληροφορικής. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για το τι προτείνεται να γίνει με τα χρήματα αυτά. Αν μου δώσετε άλλα 60 δευτερόλεπτα όμως, θα σας εξηγήσω το εξή. Πού μπορούμε να γίνουν μικρέ και ωραίε περικοπέ. Υπάρχει ένα κοιώσιο που μπορεί κανείς να αγοράσει εφημερίδες στο ισόγειο του Κοινοβουλίου. Για πολλά χρόνια αναρωτιέμαι. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι και παίρνουν μια στίβα εφημερίδες και μετά απλώς υπογράφουν. Και εγώ ρώτησα τι γίνεται, πώς γίνεται αυτό και μου είπε ο υπάλληλο ότι αυτό είναι για τις πολιτικές ομάδες. Λυπάμαι κύριε Βάλλη. η δική σας ομάδα είχε πάρει πέντε Ιταλικές εφημερίδες και δύο Αγγλικές και κάτι Γαλλικές. Τι χρειάζεστε όλες αυτές τις εφημερίδες. Έκανα ένα γρήγορο υπολογισμό. Αν έχουμε 7 ομάδες, μπορούμε να εξοικονομήσουμε 28.000 το χρόνο, αν δεν δίδονται δωρεάν όλες αυτές οι εφημερίδες. Ευχαριστώ. Έχετε δικαίωμα να απαντήσετε κύριε Βάλλη. Ευχαριστώ. Αυτές οι μικρές οικονομίες που μπορούν να γίνουν μπορούμε να τις δούμε γύρω από ένα τραπέζι σε επίπεδο όλων των ομάδων. Είδα ομπρέλες, κάποιος μου είπε για φρίσμπι, για μπαλόνια, μπάλες. Όλα αυτά είναι δαπάνες έξοδα που πάντα γίνονταν. Μπορούμε να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, να τα δούμε όλα αυτά τα τα έξοδα. Και κατά την άποψή μου θα φτάναμε και τις δεκάδες ε, ευρώ. Πρέπει να δούμε το καθένα έξοδο ξεχωριστά. Ε, τα μικρά έξοδα μπορεί να δώσουν τα μεγάλα αποτελέσματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και είναι δίκαιο σε κάποιες περιπτώσεις να αυξηθεί ο προπολογισμό λόγω χάρη για τους βοηθούς. Έχει πολλέ ευθύνε ο ρόλο του. και η δική μας ιδιότητα. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε του πόρου, εξορθολογίζοντας τι δαπάνε και όχι αναγκαστικά αυξάνοντα. Αυτό γίνεται σε πολλέ περιπτώσει στα κάτι μέλη, σε αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση, σε μικρά ή μικρότερες αρχές, σε επίπεδο περιφερειακό ή επαρχιακό. Πρέπει να το κάνουν και τα μεγάλα θεσμικά όργανα όπως το κοινοβούλιο. Η μισθή κάποιε φορέ είναι διεγκωμένη και αυτό πρέπει να το δούμε ή τα έξοδα των ομάδων, οι συνεισφορές στα κόμματα και τα ιδρύματα. Κάποιες φορές ενισχύονται και από εθνικές συνεισφορές. Εδώ έχουμε εκατομμύρια ευρώ. Εδώ πρέπει να μπει ένα όριο. Ας συναντηθούμε λοιπόν και ας ε, τα μελετήσουμε μαζί. Ο λόγος στον κύριο Ντεπρέ για να ολοκληρώσει. Αναγνωρίζουμε νομίζω όλοι Στην στη δική του κατηγορία ο καθένας και 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν μια προσπάθεια ελέγχου των δημοσιονομικών τους για να μειώσουν το έλλειμμα και να συγκρατήσουν την, το χρέος, το ποσοστό χρέωσης. Θέλουμε επενδύσεις και κινητοποίηση των ε, οικονομιών των δαπανών, των ιδιωτών, συγγνώμη, με το πρόγραμμα Juncker και το Στρατηγικό Ταμείο Επενδύσεων. Η αρχή τώρα του προπολογισμού βασίζεται, η δημοσιονομική αρχή της Ένωσης βασίζεται στο παράδειγμα που δίνει το Κοινοβούλιο ε, και πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί για να υπάρχει συνολικά έλεγχος των δημοσιονομικών. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να παίρνει την ελευθερία να μην είναι παράδειγμα ορθολογισμού και ελέγχου ε, εσόδων-εξόδων για να υπάρχουν καλές επιδόσεις. Κύριε Ντεπρέ, κύριε Ντεπρέ, με τις βαλικές αρχές θα έχετε και μια διαμεσολαβητική δράση για να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε στην έδρα του Κοινοβουλίου να πετύχουμε κάποια πράγματα. Κύριε Ντεπρέ, κύριε Πρόεδρε, για αυτό το τελευταίο σημείο επιφύλαξη, διότι εξ όσων γνωρίζω το Προεδρείο είναι υπεύθυνο για αυτό το θέμα. Με τιμάτε λοιπόν, αλλά δεν είμαι ακόμα μέλος του Προεδρείου. Νομίζω θα το ε, αναλάβει αυτό το Προεδρείο με όλο του τα μέλη και εγώ δυστυχώ δεν είμαι ένα από αυτά. Πρόεδρο, θα αποσύρω αυτό που είπα. Ε, λοιπόν, κάτι που είπα, ο προπολογισμό του 2016 γνωρίσε και πολλού άλλου προπολογισμού προηγουμένω. Δεν ήταν λοιπόν παρθενά έδαφο αυτό για μένα. Υπήρχαν πολλά που ήδη είχαν αποφασιστεί προηγουμένω. Και είναι ενδιαφέρον να σας πω για την εξέλιξη κάποιων κατηγοριών ε, δημοσιονομικών δαπανών του Ευρωκοινοβουλίου από το 2009. Και δεν τα είχα αναλάβει εγώ γιατί δεν ήμουν εδώ. Αλλά κάποιοι από εσά είσαστε εδώ τότε. Πρώτο σημείο. Ε, τα κονδύλια για τα κόμματα και τα ευρωπαϊκά ιδρύματα. Από το 2009 ε, μέχρι το 2014 167%. 167% αύξηση. δύο Σε ό,τι αφορά δαπάνες των μελών, μισθούς, συντάξεις, έξοδα μετακίνησης, 31% αύξηση. Βοηθή, συν 25% από το 2009 στο 2015 δηλαδή λιγότερα για τους βοηθούς από το μέσο όρο της γενικής αύξησης των εξόδων του Κοινοβουλίου που ήταν 26% ο μέσος όρος. Οι αριθμοί τώρα είναι, δεν το λέω εγώ, τα αποτελέσματα αυτά είναι αποτελέσματα αποφάσεων που ελήφθησαν μεταξύ 2009 και 2015. Οπότε εργάζομαι ε, με αυτά τα στοιχεία και το έχω μπροστά μου. Άρα εκεί που θέλετε να κάνω τις μεγαλύτερες περικοπές θα πρέπει να είναι στα κόμματα και τα ιδρύματα. Και θα ήθελα πολύ να δω και τι απόψει όσων είναι εδώ γύρω από το και θα έρθουν γύρω από το τραπέζι, αλλά και οι δαπάνε των ε, μελών, που ξεπερνούν το μέσο όρο των ε, μελών, τον όρο των ε, εξόδων. Εσεί πρέπει να αποφασίσετε, δεν τα φαντάζομαι αυτά. Για τι οικονομίε μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ξέρετε ότι καταργήσαμε το σερβίρισμα καφέ. Ή μπορούμε να καταργήσουμε και το ζεστό νερό στα ντου. Ποιο κάνει ντου. Εδώ. Μπορούμε να τα πουλήσουμε τα ντους. Μπορεί να φέρνει κανείς και χαρτί υγεία στις τουαλέτες. Ε, συμβαίνει σε κάποιες χώρες όπως τις Αφρικανικές. Δεν υπάρχουν όρια στην οικονομική πολιτική. Απλώς πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα κάνουμε τις ευφιέστερες επιλογές. Και να έρθω στο ύψος των οικονομιών. 10 εκατομμύρια οικονομία μας ζητούνται από το Γενικό Γραμματέα βάσει της συμβαστικής της τελευταίας συνεδρίασης. Ψεύδος 10 εκατομμύρια οικονομίες επιπλέον διότι η αύξηση των σχετικών δαπανών για τους υπαλλήλους και το σύνολο των εργαζομένων στο Κοινοβούλιο είναι 2,8% το 2016, εάν λάβει κανείς υπόψη την τιμαρρύθμιση και την ε, αύξηση προβλέπεται από τον ιστορικό κανονισμό μια πρώτη αύξηση τον Ιούλιο φέτος με 2% και 1,8% από τον Ιούλιο του 2016. Δηλαδή συνολικά για το 2015 1,5% ε, συν τα ετήσια συν όσα ορίζονται από το καταστατικό. Από τον κανονισμό. Θα έχουμε 2,8% αύξηση λοιπόν σε ένα δις ε, δαπάνες στο κοινοβουλίου. Όταν λέμε λοιπόν ότι η αύξηση είναι 1,6% κατά μέσο όρο, στα 1 δις 11 θα πρέπει να βρούμε και τα 11 που μας λείπουν. Άρα στα 10 εκατομμύρια δεν είναι 10 εκατομμύρια οικονομίες, είναι 21. Και για κάποιες συγκεκριμένε ερωτήσεις στην πρώτη ερώτηση του κυρίου Γκάγκερ. Θα σα απαντήσω και στι τρει ερωτήσει σα, κύριε Γκάγκερ, υπάρχουν και άλλε. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε πρόεδρο. Ο κύριο Γκάγκερ νομίζω έχει μια συμπληρωματική παρατήρηση, όχι. Ναι, ναι. Εγώ θα αφήσω τον κύριο Ντεπρέ αν προτιμάει να μιλήσει ω το τέλος. Υπάρχει το 31% το οποίο υπολογίσατε, το 1,3% έχει να κάνει με, το, την εφαρμογή του νέου καθεστώτος των βουλευτών που ξεκίνησε το 2009. Είμαστε σε μια δημόσια συνεδρίαση που περνάει και στο διαδίκτυο. Όταν λέτε ότι αν πείτε καλύτερα τα ποσά τα οποία είναι στη διάθεση των βουλευτών ανεβαίνουν κατά 30% αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε ορισμένους. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με το νέο καταστατικό των βουλευτών που τέθηκε σε εφαρμογή το 2009 και ίσως όλα αυτά έχουν να κάνουν και με, το, με τα ποσά τα οποία αφορούν την ε, αποχώρηση βουλευτών και τα κτλ. Ευχαριστούμε, αλλά απλώς επιβεβαιώνεται αυτά που είπα πριν, δηλαδή ότι υπάρχουν δαπάνες όπως του βουλευτικού καθεστώτος και την, την αριθμική αναπροσαρμογή που δεν μπορούν να μειωθούν. Δεν μπορούμε να τις μειώσουμε. Και άρα πρέπει να μειώσουμε από άλλα. Τώρα, άλλα ερωτήματα. Τα 15 εκατομμύρια είπα ότι είναι πρόταση του Γενικού Γραμματέα, την οποία δεχτήκαμε όλη τη διαφορά μεταξύ τρεχουσών δαπανών και εξαιρετικών του 16. Αυτός ο αριθμός των 15 εκατομμυρίων προτάθηκε από τον Γενικό Γραμματέα και το θεωρήσαμε maximum και είπαμε ότι το ακριβές ποσό θα καθοριστεί με βάση συγκεκριμένε προτάσεις που θα μας κάνει. Ας πούμε πόσα για τα τζάμια, πόσα για τα, τα νέα συστήματα ασφάλειας στις πόρτες, για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος κλπ. Λοιπόν τα 15 εκατομμύρια είναι ένα μέγιστο ποσό για την ενδυνάμωση των μέτρων ασφαλείας. Τώρα το 5% μειώνουμε κατά 5% γενικά 1% το χρόνο δηλαδή. Η πρόταση του Γενικού Γραμματέα προβλέπει αντικειμενική μείωση 57 θέσεων συν 2 σε συμφωνία με την αρμόδια επιτροπή. 59 ε, θέσεων δηλαδή ακριβώς το 1%. Αλλά ο Γενικός Γραμματεύς λέει ότι πρώτον αν θέλουμε να ενδυναμώσουμε την ασφάλεια, τότε χρειάζονται όχι μόνο εγκαταστάσεις αλλά και προσωπικό. Πρέπει να ενδυναμωθούν ορισμένες ομάδες φυλάκων, άρα πρόσθετα έξοδα. 27 πρόσωπα είπε ότι χρειάζονται παραπάνω. Και ρωτήσαμε, ζητήσαμε ενδυνάμωση και της γραμματείας των επιτροπών για καλύτερο έλεγχο για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και την καλή χρήση του προϋπολογισμού. Ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν εδώ πρότεινε 20 άτομα. Διαβάζω τις τροπολογίες των ομάδων, οι οποίες λένε καλά να ενδυναμωθεί η γραμματεία των επιτροπών, αλλά εσωτερικά, αναδιάρθρωση εσωτερική όχι προσλήψεις. Άρα πρέπει ο Γενικός Γραμματέας να έρθει να μας πει τι μπορεί να κάνει ως εσωτερική αναδιάρθρωση. Και αν δεν γίνεται, εμείς θα αποφασίσουμε αν δεχόμαστε ή όχι νέες προσλήψεις. Υπάρχει όμως μεγάλη διαφορά επίσης με την Κομισιόν για τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση του προσωπικού. Όταν αποφασίσαμε να δεχτούμε την διεθνοποίηση της ασφάλειας και να μην περνάμε πια από εξωτερικά συμβόλαια θα χρειαστούν και άλλα άτομα. Και ο κύριος Πρέζα που είναι εδώ παρόν μπορεί να το επιβεβαιώσει. Πρέπει να δούμε σε τι πραγματικά βασίζονται όλα αυτά, τι πραγματική μείωση του προσωπικού μπορεί να γίνει και ποια είναι πλασματική μόνο. Άλλο ερώτημα στρατηγικής σημασίας. Τα μη χρησιμοποιούμενα κονδύλια. Για πέρυσι ξέρω ότι είναι πάνω από 60 εκατομμύρια. Τι έγινε με αυτά. Αν αναλύσουμε καλά τον προϋπολογισμό βλέπουμε ότι δεν προβλέπει δαπάνες για το κτίριο Κόνραντ Αντενάουερ στο Λουξεμβούργο, το ΚΑΝΤ. Επίσης ζητήσαμε να μας εξηγήσουν πώς χρηματοδοτείται το κτίριο Κάντα. Είναι κάτι ανάλογο, αν και πιο πολύπλοκο, με εκείνο που μας εξήγησαν για το δικαστήριο και τον καινούργιο του πύργο. Δεν προβλέπεται κανένα κονδύλιο για τη χρηματοδότηση του Κάντα. Εγώ θέλω πλήρη διαφάνεια. Πλήρη. Αλλά τότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε πόσο κοστίζει το κτίριο CAD και τι πρέπει να χρηματοδοτήσουμε το 16. Να προσθέσουμε δηλαδή 142 εκατομμύρια. Αν θέλετε, εγώ θα το κάνω. Το βάλω. Αλλιώς χρηματοδοτούνται με δύο τρόπους. Από συλλογή και από δάνεια που επιβαρύνουν και αυτά τον προϋπολογισμό. Εγώ θέλω διαφάνεια. Αν το αποφασίσετε έτσι να γίνει. Εσείς θα αποφασίσετε. 142 εκατομμύρια πρόσθετες δαπάνες για το 16 και δεν το αποφασίζω εγώ. Δεν είπα εγώ ότι οι εργασίες πρέπει να γίνουν. Τι άλλο τώρα. ξέρω ότι μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν πολλές εξοικονομήσεις, αλλά το πρόβλημα είναι λεπτό για ορισμένα θέματα, γιατί το Προεδρείο είναι αρμόδιο. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας, ας πούμε, ο κανονισμός για τους τοπικούς βοηθούς. Αυτή την αύξηση μόνο το Προεδρείο μπορεί να την αποφασίσει. Μπορούμε να το ζητήσουμε στη συμφωνία, να ληφθούν μέτρα που να μην εφαρμοστούν αν δεν τροποποιηθεί πρώτα ο κανονισμός για τους τοπικούς βοηθούς. Αλλά το Προεδρείο θα τα αποφασίσει. Οι γραπτές ερωτήσεις ας πούμε. Έχω δει πόσες είναι. Δέκα βουλευτές, δέκα, είναι υπεύθυνοι για πάνω από τις μισές γραπτές ερωτήσεις που κατατίθενται. Δέκα. Δεν θα τους ονοματίσω. Και σε τι χρησιμεύει αυτό. Απλώς και μόνο να έχουν καλή θέση σε αυτό το ηλίθιο σύστημα ranking που βάζει στην ίδια θέση κάποιον που γράφει εκθέσεις επί μήνες και μήνες και άλλον που απλώς καταθέτει με το φτιάρι γραπτές ερωτήσεις. Και εδώ το Προεδρείο. Το Προεδρείο. Το Προεδρείο πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνουμε με τις γραπτές ερωτήσεις. Έχω κάνει πρόταση στο κείμενό μου, κάνω. Ε, μου είπανε, μα μην πάτε τόσο μακριά, το Προεδρείο θα αποφασίσει. Άλλο, οι επεξηγήσεις ψήφου. Και εδώ μπορούν να γίνουν σημαντικές οικονομίες. Παραδείγματο χάρη να αποφασίσουμε ότι οι επεξηγήσεις ψήφου που γίνονται μετά την ψηφοφορία. Έχει λήξει η συζήτηση, έχει γίνει η ψηφοφορία αυτός που κάνει επεξήγηση ψήφου το κάνει για τις εκλογές του, όχι για τους συναδέλφους του που έχουν φύγει ήδη. Αν πούμε απλώς ότι δεν θα γίνεται μετάφραση, να μιλάει στη γλώσσα του, να γράφεται στη γλώσσα του, θα γίνουν σημαντικές εξοικονομήσεις για αποδιερμηνία και μετάφραση και καταγραφή. Αλλά και αυτό το Προεδρείο πρέπει να το αποφασίσει. Μου λένε μην το προτείνετε, είναι δικαιοδοσία του Προεδρείου. Ναι, αλλά μάλιστα κύριε Πρόεδρε, αλλά υπάρχουν ομάδες που συνεχώς μου λένε, μου το υπενθυμίζουν, όχι πάντα οι ίδιες, ότι δεν πρέπει να εμποδίζω και να μπαίνω στα χωράφια του Προεδρείου. Λοιπόν τώρα, ξέρω ότι οι προτάσεις μας που τις διαπραγματευόμαστε τώρα δεν είναι ιδεώδης, αλλά εγώ εξυπηρετώ απλώς την Επιτροπή Προπολογισμών. Αν μου πείτε να μειώσω αυτά που ζητάμε θα τα μειώσω, αλλά εγώ σας επαναλαμβάνω δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να ζητήσουμε από το Προεδρείο να δεχτεί πάνω από 22 εκατομμύρια μειώσεις εξοικονομήσεις. Τα 10 εκατομμύρια δηλαδή που θα προτείνει ο Γενικός Γραμματεύς και τα 12 που σημαίνουν τις αλλαγές στο προσωπικό. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά μας. Πιστεύω ότι πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής στην ε, διάβια και την οξυδέρκεια των παρατηρήσεών σας και την ε, απόλυτη επαγρύπνηση που έχετε για τα θέματα αυτά. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με απόλυτη διαφάνεια. Αυτό πρέπει να σημαίνει η λιτότητα του υπολογισμού για τις ε, λειτουργικές δαπάνες της επενδύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να δείξουμε κάποια ευφυΐα στα θέματα αυτά όπως λέτε κύριε Ντεπρέ για να μπορούμε να είμαστε και κατανοητοί. Μπορούμε να παραμείνουμε λοιπόν σε αυτό το επίπεδο. Κύριε Τάραν, θέλετε να πείτε κάτι. 30 δευτερόλεπτα, εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή αυτά που είπε για τις επεξηγήσεις ψήφου. Αλλά θυμάμαι ότι ήμουνα στην Ολομέλεια σε κάποια συζήτηση για την σήμανση των προϊόντων κρέατος και κάποιος ε, Σκοτσέζος μίλησε για το Ρόμπερτ Μπέρνς και το Χάγκης και αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ όμορφο. Πολύ ωραία λέει ο και εγώ όταν ήλθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εντυπωσιάστηκα που οι υπεξηγήσει ψήφου γίνονται μετά την ψηφοφορία. Γιατί κανονικά σε ένα κοινοβούλιο προσπαθεί να πείσει κανεί του συναδέλφου του πριν να λάβουν μια απόφαση. Το να εξηγεί κανεί τη θέση του μετά από την απόφαση, ναι, εντάξει, αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιε εξοικονομήσει. Όπω το προτείνει ο κύριο Ντεπρέ και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασιστεί και από το Προεδρείο. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά εκεί όπου βρίσκεται η πεμπτουσία των πολιτικών ομάδων στο, στο Προεδρείο. Οι σκιώδεις οι τέσσερις είναι διάσωμα μαζί με τον κύριο Ντεπρέ το απόγευμα. Και εδώ έχουμε κάτι διάφορο, στα διάφορα. Εάν όχι, καλό Πάσχα αγαπητοί συναδέλφοι. Και μια πολύ ευχάριστη πράσινη εβδομάδα.